Ε, την ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ισχυωτικό χαρακτήρα. Πρώτος, έχει το λόγο ο εισηγητής, η εισηγήτρια μάλλον, η κυρία Ίσκρα Μιχαήλωβα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, Τα νησιά, οι νησιωτικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφοροποιούνται πλήρως από τις υπηρετικές περιφέρειες. Βάσει το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται ότι οι νησιωτικές περιοχές, το σύνολό τους, αντιμετωπίζουν μόνιμα μειονεκτήματα. Η έκτη έκθεση, λοιπόν, όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική συνοχή, Αναφέρει ρητά ότι η οικονομική κρίση επηρέασε πολλές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επηρέασε όλος ιδιαίτερος και πολύ περισσότερο τις νησιωτικές περιοχές. Τα νησιά λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Στην Ευρώπη παρατηρούνται πολλές αλλαγές ε, σήμερα, μεταξύ άλλων ε, δημογραφικές αλλαγές, ε, θέματα ενεργειακά κλπ. κλπ. Όλα αυτά είναι προκλήσεις. Και οι νότιες νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης επηρεάζονται πολύ και από το προσφυγικό. Τα φυσικά μειονεκτήματα πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη των ε, νησιών και γι' αυτό και θα έπρεπε να μπορούν τα νησιά να χρησιμοποιούν περισσότερο τις ευκαιρίες που προσφέρονται, για παράδειγμα μέσω της ψηφιακής ατζέντα. Επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα νησιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να πάρει μέτρα για να βελτιώσει τη συνοχή στις ε, νησιωτικές αυτές περιοχές. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν ετοιμάζει την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Οι νησιωτικές περιφέρειες δεν πήραν καμία ειδική χρηματοδότηση στα πλαίσια αυτού του οικονομικού προγραμματισμού. Το μόνο που τους παραχωρήθηκε ήταν η δυνατότητα διαφοροποίησης των ποσοστών συγχρηματοδότησης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν και εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων της ΔΕΚΗ θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή το εξή. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει σαφή ορισμό της μορφής που πρέπει να έχουν τα μόνιμα μειονεκτήματα, όποια και αν είναι αυτά, όπως αναφέρει το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, ποια είναι τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά τα νησιά έτσι όπως αναφέρονται στο ΝΑΤ επίπεδο 2 και 3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν τι μέτρα θα πάρει προκειμένου να αντιμετωπίσει τα μειονεκτήματα αυτά και τι δράσεις σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή στο μέλλον προκειμένου να συμμορφωθεί προς το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι όπως γνωρίζετε τα νησιά και τα φυσικά τους μειονοκτήματα πρέπει να αναγνωρίζονται. Πρέπει να αναγνωρίζονται μάλιστα ως σαν μόνιμα εμπόδια για την ε, συνοχή στα νησιά αυτά. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ρωτάω, πιστεύει ότι θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι δείκτες εκτός από το καθάριστο χώριο προϊόν, άλλοι δείκτες δηλαδή, οι οποίοι να μην έχουν να κάνουν μόνο με, την, ε, με τους οικονομικούς δείχτες, με τα οικονομικά χαρακτηριστικά, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να λυθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, αφού τα νησιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα εξαιτία των ε, μειονεκτημάτων τους και της γεωγραφικής τους θέσης. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω και προσβλέπω στην απάντησή σας. Ευχαριστώ. Και τώρα έχει το λόγο η Επίτροπος η κυρία Κρέτου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί κύριοι βουλευτές, αγαπητή κυρία Μιχαήλωβα και συνάδελφοι, καλημέρα όλοι. Να αρχίσω με τις ευχαριστίες μου προς την ε, Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής του Κοινοβουλίου για αυτή την προφορική ερώτηση που αφορά την ε, βοήθεια προς ε, τις νησιωτικές περιφέρειες μέσω των διαρθωτικών ταμείων και του Ταμείο Επενδύσεων. Έχω προβληματιστεί για την κατάσταση. Στην Γουαδελόπη κάναμε την ετήσια συνάντησή μας, αλλά και στην Ρενιό. Επίσης και στο Στασβούργο τον ε, Ιανουάριο συναντηθήκαμε με τον αρμόδιο συνάδελφο της Επιτροπής και νέα βουλευτές για αυτές τις ε, περιφέρειες ε, τις απότερης περιφέρειες με τον κύριο Βέλα συναντηθήκαμε και είπαμε για αυτήν την περίοδο 2014-2020 να δούμε τι θα γίνει και πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ε, αυτές τις περιφέρειες που βρίσκονται τόσο μακριά από την ε, Ευρώπη και έχουν επίσης συγκεκριμένα προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Όπως γνωρίζετε τα ευρωπαϊκά ταμεία έχουν μακρά παράδοση επιτυχούς υποστήριξης των περιφερειών που έχουν ε, κάποια ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά αλλά και ε, για τις νησιωτικές περιοχές ισχύει αυτό, υπάρχουν προβλήματα και σχετικά με το περιβάλλον και γενικά απαιτείται μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Κατά τη γνώμη μου, καλύπτεται το πρόγραμμα από τον ε, κανονισμό, ο οποίος αφορά την περίοδο 2014 2020. Οπότε και αυτό και θέλουμε να έχουμε κάποιες ε, συμφωνίες, εταιρικέ σχέσεις και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να εντοπίσουμε αυτά τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν αυτές οι περιοχές που έχουν καμιά φορά πάγια προβλήματα και σοβαρά προβλήματα. Ε, ήδη υπάρχουν κάποιες παρεκκλήσεις όσον αφορά τις ε, επενδύσεις και όσον αφορά τις χορηγίες του Ταμείου Περιφερειακής ανάπτυξης και οπότε εφαρμόζονται με ε, ευελιξία σχετικές διατάξεις για να καλυφθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα αυτών των περιφερειών, των νησιωτικών περιοχών που έχουν και αυτά τα νησιά κάποιες παρεκκλήσεις υπέρ τους για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τις ε, πάγιες και σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Ακριβώς όπως αναφέρατε και εσείς Νομίζω ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε περισσότερο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά ε, αυτές τις περιοχές που είναι στην κατηγορία 1 και 3 και θέλουμε να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τους ε, δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Πάντως, τα στοιχεία τα οποία έχουμε δεν χαρακτηρίζονται από αρκετή ακρίβεια για να μπορούμε να δούμε τι γίνεται σε όλες τις νησιωτικές περιφέρειες. Πάντως εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια συλλογής ε, δεδομένων ούτω ώστε να έχουμε μια καινούργια έκθεση για την ε, συνοχή και να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καλή εικόνα της κατάστασης. Ευχαριστώ και θα παρακολουθήσουμε προσοχή τη συζήτηση. Και τώρα, λέει ο Πρόεδρος, έχουμε τις παρεμβάσεις από πλευρά των πολιτικών ομάδων. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει τον λόγο ο κύριος Τσίκο. Πολύ σημαντική μέρα για μένα κύριε Πρόεδρε. Έχω την πρωτοβουλία μου ε, λόγω αυτής της ε, διαδικασίας που βλέπετε και γι' αυτό τώρα ε, έφτασε στην Ολομέλη αυτό το σημαντικό θέμα. Και θέλω τώρα να στραφώ στην Επίτροπο για να μπορέσω να τη πω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, να καταλάβουμε καλύτερα πώς είναι δυνατόν να έχουμε συγκεκριμένο προβληματισμό που να αντισχύσουν την πραγματικότητα. Διότι τα νησιά αυτά δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά. Σήμερα αυτέ οι νήσοι έχουν ε, μειονέκτημα. Και θα πρέπει επομένω να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν μπορεί να κάνει αυτή την υποστήριξη. Και θα πρέπει να αποφασιστεί αν είναι νόμιμες οι κρατικές ενισχύσεις. Γιατί έχουμε τις ε, ε, πολυεθνικές οι οποίες φεύγουν από τα νησιά. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ανταγωνιστικότητα τα νησιά. Δεν είναι δυνατόν με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα νησιά να τα καταφέρουν διότι κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει εγκατάλειψη. Οπότε θα πρέπει όταν μιλούμε για μεταφορές προσώπων ότι τι θα γίνει με το μονοπόλιο, τι θα γίνει επίσης με τον τουρισμό που δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν μπορεί να υποστηριχτεί γιατί υπάρχει εποχιακός χαρακτήρας οπότε με αυτούς τους κανονισμούς για τους οποίους μιλήσατε κυρία Επίτροπε ε, θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν επαρκούν. Θα πρέπει να ενισχυθούν γιατί οι στόχοι μας έχουν στρατηγικό χαρακτήρα. Μιλούμε για περιοχές που είναι εγκατελειμμένες. Οπότε θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί η τοποθέτησή σας και να θα πρέπει να γίνει καινούριος προγραμματισμός. Σας ευχαριστώ. Και τώρα για τους ε, σοσιαλδημοκράτες έχει τον λόγο η κυρία Τζουφρίντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την δουλειά τους σε σχέση με αυτό μας το κείμενο. Ευχαριστώ και σας που ήρθατε κυρία Επίτροπε γιατί ε, δίνετε αυτή την προσοχή ε, στις ε, νήσους. Από την Σικελία προέρχομαι και επομένως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την κατάσταση. Πρόκειται για περιοχές που έχουν πάρα πολλές αδυναμίες και διαρθρωτικές και από πλευράς ε, γεωγραφίας. Υπάρχει πλούτος αλλά υπάρχουν και πολλές αδυναμίες οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημάνει ακριβώς ποια είναι τα μειονεκτήματα να δει τι λείπει, τι εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη των νησιών της ε, Ένωσης. Δεν υπάρχει ε, κινητικότητα, τα καύσιμα κοστίζουν περισσότερο. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους και οι τουρίστες δυσκολεύονται να πάνε σε αυτά τα νησιά. Άρα χρειάζονται πόροι, χρειάζεται προγραμματισμός συγκεκριμένος να λάβει υπόψη την ιδιορυθμία των νήσων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μια ειδική ομάδα γκισέα, το πούμε, με κάποιους ειδικού και να καλύψει αυτές τις περιφέρειες. Έχουν πολλά να συμβάλλουν ε, στην ανάπτυξη νήσι όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όσον αφορά την βιολογική γεωργία. Ζητάμε επομένως έντονα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τα νησιά. Ο Πρόεδρος. Ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δεν είναι πάντα εύκολη η ζωή σε ένα νησί. Τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά τα πράγματα γιατί και εγώ σε νησί ζω. Λείπουν προϊόντα, δεν έχουμε καλές συνδέσεις, δρομολόγια, υγεία, παιδεία. Αυτές είναι ορισμένες μόνο προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες. Ούτε δουλειές υπάρχουν στα νησιά γιατί ε, έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή ο κόσμος φεύγει από τα νησιά και αυτό οξύνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα. Ωστόσο, εμείς δεν θα πρέπει να απογοητευόμαστε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, αξιοποιήσουμε το δυναμικό των νησιών μας θα πρέπει να προσελκύσουμε επενδυτές και εργαζομένους. Αυτό γίνεται μόνο με ευνοϊκή φορολογική πολιτική απορρίθμιση και επενδύσεις στις υποδομές σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου φαντάζομαι σε αυτό. Οπότε σας παρακαλώ να υποστηρίξετε τις τροπολογίες που έχω υποβάλει μαζί με τον συνάδελφο Λούαρ από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Και τώρα από τους φιλελευθέρους το λόγο έχει ο κύριος Γιάκοφσιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, τα νησιά δεν είναι μια στατιστική κατηγορία και μόνο. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με ταξινόμηση. Είναι η ζωή ίδια. Δυστυχώς όμως η ζωή είναι πάρα πολύ σκληρή και κινδυνεύει ε, να ερημώσει. Επαναλαμβάνω, δεν είναι στατιστική ε, τα νησιά ΝΑΤΣ 2, ΝΑΤΣ 3. Έχουμε πολλά μικρά νησιά στη χώρα μου, πάρα πολύ μικρά νησάκια, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει κανείς. Η Κροατία είναι μία από αυτές τις χώρες που έχουν πάρα πολλά νησιά. Και έχουμε πάρα πολλά κατοικημένα μικρά νησάκια. Και η ζωή στα νησιά, πιστέψτε με, είναι πραγματικά πάρα πολύ σκληρή σε όλες τις μορφές και τις εκφάσεις της. Θα ήθελα να σας πω τελικά ότι αν χάσουμε το νησιωτικό χαρακτήρα, την ταυτότητα των νησιών μας, θα χάσουμε ε, την ταυτότητά μας σε πολλά κράτη-μέλη. Και τελικά θα χαθεί η ίδια η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε και στα νησιά. Από την Κύριος Προπάτη Μόλις, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Κρέτσου, το άρθρο 174 παραμένει κενό γράμμα στην εφαρμογή πολιτικών που να ενισχύουν τη συνοχή στις νησιωτικές περιοχές. Και η Κομισιόν πρέπει να κάνει περισσότερα για τα νησιά της Ευρώπης και ιδιαίτερα για τα νησιά του Αιγαίου. Η Λέσβος ένα από τα ελληνικά νησιά στο αιγαίο έχει πληθυσμό 85.000. Το 2015 υποδέχθηκε 500.000 πρόσφυγες. Κάτοικοι της Λέσβου μαζί με την εθελόνδρια και γνωστή ηθοποιό Σούζαν Σάραντον έχουν προταθεί για Νόμπελ Ειρήνης γιατί σε αυτούς τους πρόσφυγες του πολέμου έδειξαν ανθρωπιά και αλληλεγγύη καλύπτοντας τα ελλείμματα της Ευρώπης. Αλλά και εσείς πρέπει να κάνετε περισσότερα ως Κομισιόν γιατί αυτά τα νησιά είναι χώροι σημαντικού τουριστικού ενδιαφέροντος με μεγάλα ελλείμματα υποδομών για τους κατοίκους, με τεράστιο κόστος μεταφορών και η εμπροστοφυλακή της Ευρώπης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος. Όχι λόγια λοιπόν μόνο, αλλά έργα. a nome del κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κυρία Επίτροπε. Ευχαριστούμε που ήρθατε για αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Σημαντικό για την Ιταλία. Εμείς συμφωνούμε με τα περισσότερα σημεία αυτού του ψηφίσματος. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν άλλα κριτήρια και όχι μόνο το ΑΕΠ. Στη Σαρδινία ας πούμε. Ε, όλα πάνε καλά λέει. Εκεί ε, είμαι στο 77% του μέσου όρου, αλλά όμως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχει μεγάλη ανεργία. Θα πρέπει να σας πούμε ότι θα πρέπει η Ένωση να προσέξει, αλλά δεν το κάνει αυτό. Όχι άλλα λόγια. Θα πρέπει να βρουν κάποιες λύσεις. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Επίσης υπάρχει πρόβλημα με τη μεταφορά, τη μεταφορά της ενέργειας. Ε, δεν έχουμε απορρόφηση των πόρων γιατί υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ανικανότητα των τοπικών αρχών. Ε, άρα αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις από τον Περλουσκόνη μέχρι τον Ρέντσι. Επίσης ε, είναι και περιοχή που πλήσεται από τους σεισμούς. Μιλάμε για μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση που χρειάζεται, χρειάζονται βιώσιμες μεταφορές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όλα αυτά τα οποία αναφέρονται για την απασχόληση και την ενέργεια στο ψήφισμα. Είναι θέμα των ε, επιλογών ε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη το ότι είναι γελίες οι συνθήκες σε σχέση με τη μεταφορά ενεργείας στα στενά της ε, Σικελίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Νταμάτο και τώρα για την ε, Ευρώπη των Εθνών της Ελευθερίας. Ο κύριος Σαλβίνη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε θα πρέπει να δείτε την πραγματικότητα σε Δενία ε, και Σικελία έχουν ανεργία πάνω από 50% φεύγουν οι νέοι είναι κάτι σαν ε, απικίες πρώτα πρώτα από το Ιταλικό κράτος και τώρα από τις Βρυξέλλες δεν υπάρχει βοήθεια κακό τους κάνουν και οπότε πρόκειται για μια πολιτική που είναι ένα ναυάγιο και ουσιαστικά ε, μιλάμε για χιλιάδες εργαζομένων που φεύγουν και επίσης έχουμε πάρα πολλά προϊόντα που έρχονται από την άλλη όχθη της ε, ε, ε, Μεσογείου και έρχονται και εγκαθίστανται εκεί είναι γελία κατάσταση επίσης των μεταφορών, μόλυνση και 80% των τρένων που κυκλοφορούν με, με ντίζελ έχουν μόνο μία γραμμή και στη Σαρδινία Επίσης, τι να πούμε για τα τρένα, γιατί και εκεί λείπει ένας αυτοκινητόδρομος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, παραβάσεις και υπάρχει μονοπόλιο επίσης όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Οπότε θέλουμε να σας ζητήσουμε από πλευρά των νησιών να τους αφήσετε ίσχους, να αφήσετε τα νησιά να κάνουν μια αυτοδιαχείριση και οι να ρυθμίσουν τα θέματα της απασχόλησης. Να μην ε, θεωρείτε ότι θα τα πάνε καλά τα νησιά με την ε, υποδοχή των ε, μεταναστών. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος και τώρα θα συγκεκριμένουμε τους υπόλοιπους ομιλητές και τώρα το λόγο έχει η κυρία Φεραγκούτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς είναι πολύ ευπρόσδεκτο αυτό το ψήφισμα και συγχαρητήρια Σαλβατόρε Τσίκου για τον νησιωτικό χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι από τη Μαγιόρκα, ξέρετε. Είναι μία από τις Βαλεαρίδες ε, νήσους, ανήκουν στην Ισπανία και εμείς εδώ και καιρό αγωνιζόμαστε να μας αναγνωρίσουν οι συνθήκες σε αυτό το νησιωτικό χαρακτήρα. Και όχι μόνο, είναι και διπλός και τριπλός. Η Μενόρκα, η Φορμεντέρα, τα πιο μικρά νησιά εκεί στις Βαλεαρίδες ε, νήσους. Έχουμε πρόβλημα στη γεωργία, στις μεταφορές, στις συνδέσεις, ε, στην υγεία, στην παιδεία και πάει λέγοντας. Άρα θα πρέπει όλα αυτά κάπως να αποζημιώνονται. Αυτό το αναγνωρίζει η συνθήκη στο άρθρο 174 και όταν κάνει λόγο και για κοινωνική συνοχή και για οικονομική και για εδαφική. Όμως όταν φτάνουμε στον προϋπολογισμό αρχίζουν οι δυσκολίες. Εδώ χειροκροτώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και την πρόταση του δικού μας ψηφίσματος και της ερώτησης να δημιουργηθεί ένα θεματολόγιο ή μια λευκή ε, βίβλος για την ανάπτυξη των νησιών και να υπάρχει ανταγωνιστικότητα σε όλους τους στρατηγικούς ε, τομείς, να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και η νήση με το υπόλοιπο υπηρετικό έδαφος. Ο κύριος Παπαδάκης, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε μια Ευρώπη όπου ο σεβασμός στην ποικιλομορφία αποτελεί βασική αρχή, δεν αρκεί απλώς να γνωρίζουμε περιοχές με μόνιμες ιδιαιτερότητες και μειονεκτήματα. Τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών είναι πολλά και πρέπει να αποτραπεί από απομόνωσή τους. Χρειάζονται στοχευμένες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να ξεπεραστούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε προβλήματα πρόσβασης σε βασικά αγαθά όπως το νερό καθώς και στη στέρηση βασικών υπηρεσιών όπως της υγειονομικής περίθαλψης έχουμε το παράδειγμα των μικρών νησιών στην ελλάδα. επίσης πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιωτικών περιοχών όπως η εκμετάλλευση ποικίλων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. η μη ένταξη αυτών των περιοχών κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 14-20 θα αποτελέσει χαμένη ευκαιρία για σωστές και στοχευμένες επενδύσεις. Τέλος, να σημειώσω πως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός της Eurostat αφού η μονέοπλευρη προσέγγιση που υπάρχει με τη χρήση ενός και μόνο κριτηρίου του κατά πόσο μια νησιωτική περιοχή είναι νησιωτικό κράτος ή μη δεν δίνει βαρύτητα σε άλλα σημαντικά ζητήματα όπως το πληθυσμιακό και την απόσταση της νησιωτικής περιοχής από την υπηρετική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κύριε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, μιλώντας σήμερα για νησιωτικότητα, δηλαδή για την ανάγκη πολύπλευρης στήριξης των ευρωπαϊκών νησιών, τουλάχιστον για τη δική μου χώρα για τα ελληνικά δηλαδή νησιά δεν υφίσταται έχει καταργηθεί στην πράξη. έχει καταργηθεί πρώτον διότι και τα ελληνικά νησιά πληρώνουν τις συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών των πολιτικών της λιτότητας καταργήθηκαν ειδικά φορολογικά καθεστώτα που λαμβάνονται σε άλλα ευρωπαϊκά νησιά όπως μειωμένο ΦΠΑ προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαιτερότητες που γνωρίζουμε πως έχουν τα ελληνικά νησιά. δεύτερο ξεπουλήθηκαν τα αεροδρόμια σε ιδιωτικά και ξένα συμφέροντα με συνέπεια να αμφισβητείται αν θα μπορέσει να επέλθει μείωση του κόστους των μεταφορών που ξέρετε ότι είναι κρίσιμο όσο αφορά τα μεταφορά στα νησιά. Και τέλος υφίστανται τις συνέπειες της πολύπλευρης προσφυγικής κρίσης ιδιαίτερα τα νησιά του Αιγαίου και της ανύπαρτης ευρωπαϊκής πολιτικής αλληλεγγύης. Θα εκτιμούσα λοιπόν με την ευκαιρία αυτή κυρία Επίτροπε αν μου δίνατε μια απάντηση σε ένα ερώτημα που σας έχω υποβάλει εδώ και τέσσερις μήνες σχετικά με το τι ειδικά μέτρα παίρνετε στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής στα πλαίσια της νησιωτικότητας για τα ελληνικά νησιά που υφίστανται σήμερα που δέχονται το μεγαλύτερο προσφυγικό βάρος και στη διαχείριση των ανθρώπων και στην καταγραφή των προσφύγων και στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. σας ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ κύριε οι οποίοι ε, έφεραν στην Ολομέλη αυτή την συζήτηση και ευχαριστούμε που ήρθε και η κυρία Επίτροφο που ζητήσαμε. Κοιτάξτε, σήμερα έχουν περιθωριοποιηθεί τα νησιά και δεν είναι αυτό μόνο γεωγραφικό, είναι και οικονομικό και κοινωνικό. Τώρα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει κάποιες δράσεις για αυτή την ε, απομακρυσμένη περιφέρεια. Όμως δεν ε, υπάρχουν όλα αυτά. Είναι στο περιθώριο τα νησιά. Τι θα κάνετε για να βοηθήσετε τον, να έχουμε συμπερίληψη των νησιών στην ανάπτυξη. Θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερος προγραμματισμός για να μπορέσουν να ξεπραστούν τα προβλήματα από την νησιωτικό χαρακτήρα γιατί δεν έχουν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Εγώ παίρνω τρία αεροπλάνα για να έρθω εδώ γιατί ε, είναι πολύ μακριά και βέβαια ε, πάλι καλά ε, πρέπει να τα βρω από την τσέπη με αυτά τα έξοδα για τα τρία πλάνα. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε την περιθωριοποίηση και πώς θα υπάρχει προσβασιμότητα στις αγορές από τα νησιά. Ε, ευχαριστούμε κύριε Λαδία. Και τώρα η διαδικασία catch the ποιο ελκύει στην προσοχή του Προέδρου. Υπάρχουν πάρα πολλοί, γιατί πάρα πολύ ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα των νησιών. Και παρακαλώ, εάν θέλετε, να λάβετε όλοι το λόγο. Αλλά αυτό το οποίο επιβάλλεται είναι οι αγορητέ να λάβουν το λόγο μόνο για ένα λεπτό. Αλλιώ θα είμαι υποχρεωμένο να σα πάρω το μικρόφωνο. Κύριε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Σίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωτοβουλία αυτή. Εγώ προέρχομαι από χώρα που έχει χίλια νησιά και πρέπει να πω ότι φοβούμε για το τι θα συμβεί με τα νησιά μας. Ο κόσμος εγκαταλείπει τα νησιά, οι κάτοικοι. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο πρέπει να αναπτύξουμε καλύτερες πολιτικές. Πολιτικές οι οποίες θα έχουν ω στόχο να ενισχύσουν οικονομικά προγράμματα στα νησιά. Σήμερα βλέπουμε ότι μόνο με προγράμματα υψηλής χρηματοδότησης μέσω της πολιτικής συνοχής λαμβάνουν χώρα. Γιατί να μην είναι πιο ευέλικτη η κρατική επιδότηση όταν πρόκειται για νησιά. Γιατί να μην μπορούμε να συγχρηματοδοτήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία ταξινομούνται τα νησιά. Έτσι θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης ε, στα νησιά, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για να παραμείνει ο κόσμος στα νησιά του. Ευχαριστούμε. Πίκολα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, υπάρχουν ε, πολλά ζητήματα για τους κατοίκους των νησιών. Το ΕΠ είναι χαμηλότερο κατά 5%. Οι κάτοικοι φεύγουν από τα νησιά, δεν υπάρχουν καλές μεταφορές, ούτε καλές υπηρεσίες υγείας. Το καθάριστο χώριο προϊόν δεν είναι το καταλληλότερο κριτήριο, γιατί δεν λαμβάνονται έτσι υπόψη άλλα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τους κατοίκους των νησιών. Μιλάμε για διαφορετικούς ορισμούς. Εγώ όμως πιστεύω ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά για τα ευρωπαϊκά νησιά, κυρίως όσον αφορά τη συμμόρφωση προς το άρθρο 174 της συνθήκης οι ευρωπαϊκές πολιτικές ε, δεν έχουν, δεν είναι ποτέ οι κατάλληλες. Είμαι από την Κροατία και ζητάω, κάνω έκκληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση του κόστου ζωής στα νησιά και να προσαρμόσει την οικονομική στήριξη και τα οικονομικά προγράμματα βασί τέτοια ανάλυση. Πρέπει να βοηθήσουμε τα νησιά και να βοηθήσουμε τους κατοίκους τους να χρησιμοποιήσουν πλήρω τις δυνατότητες που έχουν. Το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ότι οι νησιωτικέ περιοχές στο σύνολό του αντιμετωπίζουν μόνιμα μειονεκτήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. τα μειονεκτήματα αυτά έχουν σχέση με τη δημογραφική τους κατάσταση αλλά και τη φυσική τους θέση. αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα νησιά να αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητα αλλά και κοινωνική συνοχή. στην ελλάδα τα νησιά αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ευάλωτα στην οικονομική κρίση αντί όμως να τύχουν στήριξης η τρόικα κατάργησε το ειδικό φορολογικό καθεστώς των νησιών του αιγαίου και αύξησε το ΦΠΑ από 13% στο. 23%. επίσης η τρόικα δρομολόγησε το ξεπούλημα στη fraport των πιο σημαντικών νησιωτικών περιφερειακών αεροδρομίων. επιπλέον τα νησιά του αιγαίου πλήττονται πλέον από τις τεράστιες προσφυγικές ροές καθώς πάνω από 600.000 πρόσφυγες φιλοξενήθηκαν σε πρώτη φάση στα νησιά του αιγαίου το 2015. Όμω η έλευση αυτού του τεράστιου αριθμού προσφύγων και η έλλειψη ε, υποδομών δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα και έπληξαν την τουριστική εικόνα των νησιών. απαιτούνται λοιπόν μέτρα συγκεκριμένα για τα νησιά του αιγαίου και κατάργηση του ΦΠΑ από το 23% μείωση τουλάχιστον στο 13%. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, εγώ είμαι από μια χώρα που έχει δύο αυτόνομες περιφέρειες στη μέση του Ατλαντικού. Μαδέρα και Αζόρες στην ε, Πορτογαλία. Οι Αζόρες είναι εννιά νησιά. Είναι ε, αρχιπέλαγος. Είναι διπλή η νησιωτικότητα εκεί. Ε, υπάρχει πρόβλημα ε, και με τους μετανάστες. Ε, δηλαδή φεύγει ο κόσμος, μεταναστεύει από Δημή στον Καναδά και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Καμιά φορά χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να πάνε από τον Καναδά ε, ή τις Ηνωμένε Πολιτείε σε ένα νησί των Αζωρών από ότι να πάνε σε ένα άλλο νησί ε, στο ίδιο αρχιπέλαγος. Είναι πανάκριβες οι μεταφορές, είναι άγωνη γραμμή και για να φτάσετε στην υπηρετική Πορτογαλία κοστίζει μια περιουσία. Εγώ κάλεσα δύο σχολεία πέρσι και μερικά παιδιά χρειάστηκε να πάρουν τέσσερα αεροπλάνα για να φτάσουν στις Βρυξέλλες. Παρακαλώ, τέσσερα αεροπλάνα. Βοηθήστε ε, τους κατοίκους ε, των νησιών αυτών, των Αζωρών και της Μαδέρας. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συνοχή και χωρίς ε, κυκλοφορία ελεύθερη των ανθρώπων αυτών. Ευχαριστώ. Ε, Ο πληθυσμός στην Ευρώπη υποφέρει από τις πολιτικές λιτότητας και τα συμφέροντα μεγάλων οικονομικών ομάδων. Τα νησιά τιμωρούνται περισσότερο, γιατί είναι εκείνα που ξεκινούν με μειονεκτήματα, έτσι κι όσον αφορά την οικονομία. Έχουμε τη Μαδέρα και τις Αζόρες, που διπλά υποφέρουν επειδή είναι νησιά, αλλά και επειδή υπάρχει το πρόγραμμα λιτότητας της Τρόικα. Οι Αζόρες και η Μαδέρα. Ο πληθυσμό εκεί κατάφερε να επιζήσει μέσα σε αυτό τον κόσμο τον φιλελευθερωποιημένο. Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πρέπει να πάει εκεί και να δει και να φροντίσουμε να υπάρξει ένα έτος για τα νησιά. Η εδαφική συνοχή απαιτεί σαφείς πολιτικές στήριξης υπέρ της παραγωγής, υπέρ των μεταφορών, προκειμένου οι κάτοικοι των νησιών να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες όπως έχουν και οι υπόλοιποι στην Ευρώπη. Ο κ. Κρυστοφόρου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρωτίστως Οφείλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό συνάδελφο τον Σαλβατόρ Τσίκου και να του δώσω τα συγχαρητήρια καθώ και στου άλλου συναδέλφου που πραγματικά άγγιξαν το ζήτημα των νησιών μα. Ευρώπη είναι και τα νησιά μα. Πρωτίστω είναι τα νησιά μα. Φανταστήκατε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και μια Ευρώπη χωρί τα νησιά. Αλλά πιστεύω ότι είναι η εποχή που πρέπει να τερματιστούν τα λόγια και να αρχίσουν οι πράξει. Τα νησιά είναι απομονωμένοι και τα αναγνωρίζουν όλα. Πιστεύω ότι συγκεκριμένα τα νησιά πρέπει να βγουν από την απομόνωση έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. πρέπει να γίνει ένα αντίστοιχο πακέτο όπως ήταν το πακέτο των Τελόρ, πακέτο Γιούγκερ, ειδικά για τα νησιά για να στηριχθούν. Μιλούμε για απομόνωση. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την πρωτοβουλία μας για δημιουργία δωρεάν δικτύου Wi-Fi για όλα τα νησιά. Θα μπορούσαν να ενισχυθεί η στήριξη για την επικοινωνία της μεταφορές στα νησιά. Θα μπορούσαν να δώσουν κίνητρα ούτως ώστε τα νησιά να μπορούν να ανταπεξέλθουν όσον αφορά τα βασικά κοινωνικά αγαθά θα μπορούσαν αυτά τα νησιά τα οποία εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση επάξια να γίνουν πραγματικά νησιά που μπορούν να προσφέρουν αλλά και να πάρουν από αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι το δικαιούνται κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, με πολύ ενδιαφέρον συμμετέχω στη συζήτηση αυτή για τις νησιωτικές περιοχές, μια που κι εγώ είμαι από τα Κανάρια, από νησιά. Βλέπω λοιπόν ποια είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020-2030. Είναι μια τεράστια ευκαιρία προκειμένου να δώσουμε όθηση και να αποζημιώσουμε τα νησιά αυτά που είναι τόσο ευάλωτα. Πρώτον, πρέπει να δούμε την απασχόληση. Οι περιοχές αυτές υποφέρουν από πολύ ψηλή ανεργία. Πρέπει λοιπόν να τις βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε το εργατικό δυναμικό, το τοπικό, ώστε να βρούνε δουλειά και να δώσουν με τη σειρά τους όθηση στην οικονομία. Πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί το κριτήριο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ως μόνο κριτήριο για την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών αυτών γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τις ενισχύσουμε οικονομικά και κοινωνικά. Πρέπει επίσης να δώσουμε όθηση στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις ε, νησιωτικές πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ. Schwab. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τη συζήτηση την παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ δεν κατάγομαι από νησιωτική περιοχή, αλλά πολλά από τα προβλήματα που ακούσαμε τα έχει και ε, η υπηρετική Ευρώπη. Υπάρχουν δυσκολίες με τη γραφειοκρατία, με τους διοικητικούς μηχανισμούς ε, που έχουν πιο δυνηρές και σκληρές συνέπειες στα νησιά και στη ζωή των ανθρώπων εκεί. Το καταλαβαίνω αυτό. Άρα θα πρέπει και τα νησιά να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τώρα η κρίση προσφυγική δείχνει πόσο σημαντικά ε, ε, είναι αυτά τα θέματα να λειτουργούν σωστά οι υποδομές στα ευρωπαϊκά νησιά. Γι' αυτό τώρα θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία που έχουμε δεδομένη της κρίσης να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να στηθούν οι μηχανισμοί, οι υποδομές, να βοηθηθούν και οι νησιώτες να ξεπεράσουν τα προβλήματα και πραγματικά και αυτό είναι ένα στοιχείο αλληλεγγύης του κέντρου της Ευρώπης και της Υπήρου ε, προς τα τα νησιά. Σόρου. Είναι σημαντική η σημερινή πρωτοβουλία από την ε, περιφερειακή πολιτική και έτσι να μπορούμε να συζητήσουμε τώρα με την Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Σε πάρα πολύ ε, λίγο χρόνο θέλω να πω το εξή μήνυμα, κύριε Επίτροπη. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την συνοχή. Αυτό το οποίο σήμερα το πρωί. για Να θυμηθούμε ότι έχουμε την πρόσφατη κρίση αυτή, η οποία χτύπησε πάρα πολύ τα νησιά και επομένω υπάρχουν και μεγάλε δυσκολίε. Υπάρχει δυσκολία όσον αφορά την ανάπτυξη. Δεν μπορούν να φτάσουν την ανάπτυξη ούτω ώστε να ε, μπορέσουν να, να μπουν στην ε, Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνοχή. Επίση σα ε, τονίζω ότι σήμερα θα πρέπει να υπάρξει ένα δίκτυο ούτω ώστε να ξεπεραστούν δυσκολίε από τα νησιά ή θα χρειάζεται συγκεκριμένη πρωτοβουλία και πρέπει κάτι να γίνει επίσης και με την ε, ψηφιακή πολιτική. Η Σικελία και η Σαρδινία έχουν πρόβλημα, πρόβλημα και με το φυσικό αέριο, υπάρχει πρόβλημα με τις ε, μεταφορές. Θα πρέπει αυτά όλα να τα, τα σιγουρέψετε για τα νησιά. Χρειάζεται κινητικότητα. Ό,τι κάνετε να το κάνετε γρήγορα, Επίτροπε. Κύριε Μπρέσο. Από την ε, συζήτηση και από όσα άκουσα προκύπτει το εξής κύριε Επίτροπε ότι τα νησιά από τη μια πλευρά έχουν κάποια στοιχεία κοινά. Όλα τα νησιά έχουν σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την υπηρετική Ευρώπη αλλά υπάρχουν και διαφοροποίησεις από το νησί στο άλλο ανάλογα με την απόσταση από την εδώ χώρα, ανάλογα με το μέγεθό του, όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτό που θέλω να σα συζητήσω είναι το εξή. Άκουσα όλα αυτά τα προβλήματα και θα πρέπει να υπάρχει μια λευκή βίβλος όπου να καταγράφονται όλες αυτές οι διαφορές, τι γίνεται με τα μεγάλα νησιά, τι γίνεται με τα μικρά νησιά, εκεί που υπάρχει πρόβλημα με τον νησιωτικό χαρακτήρα, όταν πρόκειται ας πούμε για ένα αρχιπέλαγος, τι γίνεται ε, με τα νησιά βρίσκονται στην ε, περιφέρεια ε, όπου εκείνα τα νησιά έχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Παρακαλώ να το λάβετε αυτό υπόψη. Γραπίνη. Κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ακόμα και αν δεν ζω εγώ σε νησί, όπως είπε και ο κύριος Φαπ κατανοώ πάρα πολύ καλά τα προβλήματα των νησιών τελικά είναι αντίστοιχα και με εκείνα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προάγει τις πολιτικές συνοχής έτσι ώστε να συγκλίνει το βιωτικό επίπεδο με την υπόλοιπη Ευρώπη. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που συμμετέχετε σήμερα στη συζήτηση και θα ήθελα να ε, κοιτάξετε και άλλους δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης, όχι μόνο τους οικονομικούς. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να βοηθάει τον κόσμο να αναπτύσσεται, να βελτιώνει τη ζωή του. Χρειαζόμαστε νέους δείκτες και να μην ξεχνάμε την πολιτική συνοχή στην Ανατολική Ευρώπη, όχι μόνο στα νησιά, γιατί έχουμε επαναλαμβάνω αντίστοιχα προβλήματα. Επίσης, πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορούν να απορροφούν τα κονδύλια αυτά. Ευχαριστώ. Non sono mancate le sollecitazioni, anche gli interventi forti. Ora tocca alla Commissione. Πάρα πολύ ζήτησαν λόγο και τώρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σε ερωτήσεις που υπευλήθησαν από το Ευικύκλιο. Κύριε Κρέτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στη συζήτηση αυτή. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ευθύ εξ αρχής όσον αφορά τη σημασία που αποδίδω εγώ στα ειδικά χαρακτηριστικά και τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά και οι περιφερειακές περιοχές. Όπως έχω ξαναπεί, πέρυσι συμμετείχα στην συνάντηση για τη Γουαδαλούπη φέτος η αντίστοιχη συνάντηση θα λάβει χώρα στη Μαδέρα. Πριν από δύο εβδομάδες στο Στρασβούργο συναντήθηκα με πολλούς από εσά. Συναντήθηκα δηλαδή με πολλούς ευρωβουλευτές που έρχονται από τις άκρος ε, περιφερειακές περιοχές. Ξέρω ότι θέματα που σας απασχολούν είναι οι κλιματικές αλλαγές, το ξέρω από τον κύριο Βέλα. Ξέρω επίσης ότι πολλοί από εσά αντιμετωπίζουν και ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αλία, με την ε, πολιτική μας, την αυτιλιακή κλπ. Αυτές λοιπόν οι άκρος περιφερειακές περιοχές και η νήση γενικότερα ε, φυσικά είναι μέρος των κρατών μελών. Χαίρομαι λοιπόν που το Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποχρέωσε τις χώρες μέλη να λάβουν υπόψη τους τις άκρος περιοχές στα πλαίσια των ε, αφαρμοστικών προγραμμάτων και να λάβουν υπόψη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών να είσαστε σίγουροι ότι είμαστε σε συνεχή διάλογο με τις χώρες μέλη προκειμένου να δώσουμε την προσοχή που χρειάζεται στις νησιωτικές περιοχές και τις άκρος περιφερειακές περιοχές. Σε περιοχές δηλαδή που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως ε, είπα, το πλαίσιο του Ταμείου του Επενδυτικού για το 2014-2020 είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες αυτές των νησιών. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν για το ότι έχω δώσει συστάσεις τους ε, στις αρχές των νησιών αυτών για να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Δεν φτάνει να πηγαίνει δυο φορές το χρόνο η Επιτροπή στα νησιά. Όπως λέγατε και εσείς, δεν γνωρίζουμε έτσι την πραγματικότητα. Χρειάζεται ένα συνεχής διάλογος. Μόνο με ένα τέτοιο διάλογο θα γνωρίσουμε τα ακριβή προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά. Μπορείτε να βασιστείτε λοιπόν σε μένα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ελλάδα πιο συγκεκριμένα γνωρίζετε ότι πέρυσι ζήτησα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπιστεί μια έκτακτη κατάσταση εκεί. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι καταφέραμε να αλλάξουμε τη ρύθμιση προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση 100% νομίζω ότι έτσι κάναμε ό,τι ήταν στο χέρι μας για την Ελλάδα. Συμφωνώ με τόσα είπατε εδώ. Πάνω από 180.000 άνθρωποι έφτασαν μέσα στο 2015 μόνο στην Ελλάδα. Είναι τεράστιο το βάρος αυτό για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να στηρίξει τη χώρα και προκειμένου να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Αλλά το θέμα έχει να κάνει και με την διοικητική ικανότητα. Αναφερθήκατε στη Λέσβο. Εγώ συναντήθηκα με την ε, κεφαλή του νησιού, με τις αρχές. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν χρησιμοποίησε τα ευρωπαϊκά ταμεία για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της μετανάστευσης. Υπάρχουν δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά όμως για να φτιαχτούν κινητά, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία κτλ. Η Ιταλία από την άλλη ζήτησε τη στήριξη των ταμείων αυτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει μεταφέρει σημαντικά ποσά προς την Ιταλία. Γνωρίζω τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και θέλω εδώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αντιμετωπίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες αδυναμίες των νησιών. Βλέπετε, μερικές χώρες δυστυχώ δεν επιθυμούν να εξετάζονται τα νησιά σαν μια χωρί στην περίπτωση η Ελλάδα, παρά τη, στη συνθήκη προσχώρησης ζήτησε να θεωρηθεί σαν ενιαία χώρα. Σαν μια ενιαία κατάσταση δηλαδή να επικρατήσει ολόκληρη τη χώρα. Και να μην αντιμετωπίζονται, να μην θεωρούμε ότι τα νησιά πρέπει να βρίσκονται υπό ειδικέ συνθήκες. άλλε χώρε, για παράδειγμα στην ε, Συμφωνία προσχώρηση είπε ότι η Ρεουνιόν, και Γουαδελούπη κτλ. έχουν ανάγκη από ειδικέ πολιτικές. Άρα λοιπόν είναι θέμα επιμερισμένης ευθύνης. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό είναι ευθύνη 100% των χωρών μελών. Όπως είπα ήδη, Υπάρχουν ειδικά μέσα, ειδικέ παρεκκλήσεις που χρησιμοποιούνται. Τώρα αυτό που είναι σημαντικό για την επόμενη περίοδο είναι να βελτιωθεί η περιφερειακή πολιτική για να τα αποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες όλων των περιοχών και να προλάβουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Να ξέρετε ότι είμαι στη διάθεσή σας. Ελπίζω να πετύχουμε φέτος να οργανώσουμε στις Βρυξέλλες μία συνάντηση για αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι οι νησιωτικές περιφέρειες θα μπορούν να αντιμετωπίσουν και τις σημερινές προκλήσεις και τις μελλοντικέ και να μπορέσουν να συνεισφέρουν όσο γίνεται περισσότερο στους ευρωπαϊκούς στόχους. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση των περιφερειακών περιοχών και των νήσων Ήμουνα στη Σικελία, για παράδειγμα, πρόσφατα. Θέλουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια να χρησιμοποιούνται όσο γίνεται καλύτερα, προκειμένου να υπάρχει θετικός αντίκτυπος για την οικονομία των ε, νησιών, κυρίως υπέρ της απασχόλησης. Και επίση θέλουμε να χρησιμοποιούνται όσο γίνεται καλύτερη ενεργειακή πόρη. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα που αναφέρατε, όπως επίσης και οι μεταφορές και η κακή σύνδεση. Κάποιο έλεγε ότι έπρεπε να πάρει τέσσερα αεροπλάνα για να έρθει στις Βρυξέλλες. Είναι όμως θέμα, κυριαρχίας είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητα. Η Γαλλία, για παράδειγμα, επιδοτεί από τον προπολογισμό της το κόστος μεταφοράς των πολιτών που ζουν σε αυτά τα μακρινά νησιά. Άλλες χώρες όπως η Ισπανία επίσης το κάνει. Άρα υπάρχουν χώρες οι οποίες επιδοτούν τις μεταφορές αυτές. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε όμως, γιατί δεν είναι δικό μας θέμα. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να συζητάμε τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών. Είμαι πεπισμένη ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα, ότι χρειαζόμαστε εξαιρέσεις, παρεκκλήσεις, γι' αυτό και υπάρχει επιμονή μου βάσεως συζήτηση με τους άλλους επιτρόπους στην Επιτροπή. Γιατί γνωρίζω ότι αν η ελληνική πολιτική, για παράδειγμα, είναι πολύ αυστηρή, ε, χρειάζονται παρεκκλήσεις για τα νησιά, γιατί τα νησιά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Τη προγραμματική περίοδο 2010 μέχρι το 2015 ο προπολογισμό που εσείς εγκρίνατε ως συνομοθέτες είναι ένας προπολογισμό ε, που βοήθησε λίγο. Πολλά μπορούν ακόμα να γίνουν για να καταλήξουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Με καλές ιδέες, ό,τι προτάσεις υπάρχουν είναι ευπρόσδεκτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση για αυτό το σημείο που είναι τόσο επίκαιρο, έχει